ερώσω το σώμα πως ε, μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου ο πρόεδρος την Τρίτη θα υπογράψει τέσσερα νομοθετήματα τα οποία εγκρίθηκαν με την τακτική νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού. Οι τίτλοι θα δημοσιευτούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Αυτές ήταν οι ανακοινώσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Το τελικό σχέδιο